Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Πρώτα πρώτα να σας πω πρέπει να τελειώσουμε 5.30 άρα δεν έχουμε πολύ πολύ χρόνο. Να σας καλωσορίσω όλους στη συνάντηση τους προσκεκλημένους από την Ταϊβάν ιδίω, τόσοι πολλοί εδώ Καταρχά, φαντάζομαι ότι θα καταλάβετε ότι είμαι ο κύριο Είχε άλλε υποχρεώσει δεν μπορεί να έρθει εδώ, οπότε μου ζητήθηκε να προεδρεύσω εγώ. Είναι η τελευταία δημόσια ακρόαση για την περίοδο αυτή της θητείας της Επιτροπής ΙΝΤΑ και χαίρομαι που θα συζητήσουμε εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Ταϊβάν σε αυτή την τελευταία συζήτηση. Η επιλογή του θέματο αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή μα ιδίω για το θέμα των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ένωση και Ταϊουάν που είναι εντυπωσιακέ ε, από πολλέ οπτικέ. Η Ένωση υποστηρίζει την πολιτική τη μια μία για Ταϊβάν, δηλαδή δεν έχει επίσημε διπλωματικέ σχέσει με Ταϊβάν, Ωστόσο, οι διμερεί οικονομικέ μα σχέσει είναι εξαιρετικά ισχυρέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή, το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν οχταπλασιάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Ω εκ τούτου η Ταϊάν το 2017 ήταν ο 16 ο εμπορικό εταίρο τη Ένωση. Τα τελευταία χρόνια η Ένωση ήταν η κύρια πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ταϊβάν. Οι επενδύσει αυτέ κατά μέγα μέρο πήγαιναν σε τομεί υψηλή τεχνολογία και καινοτομία, που είναι ένα από τα ισχυρά στοιχεία τη Ταϊουάν. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ε, κατατάσσει την Ταϊβάν στη 15η σειρά μεταξύ 137 οικονομιών στο, στην Παγκόσμια Έκθεση ανταγωνιστικότητα που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Παρά τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία, η Ένωση και η Ταϊβάν δεν έχουν επίσημη εμπορική συμφωνία. Ούτε καν έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις ε, μπορικών διαπραγματεύσεων, επίσημε τουλάχιστον, παρότι η Ταϊβάν είναι μέλο σε μια σειρά πολυ, πολυμερή βήματα όπω ο ΠΟΕ, ε, στον οποίο ε, εντάχθηκε το 2013. στι 12 Σεπτεμβρίου του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα όπου ζητήσαμε και παραθέτω την έναρξη διαπραγματεύσεων για διμερή συμφωνία επενδύσεων με την Ταϊβάν. Στο ίδιο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο υπενθύμησε ότι η Επιτροπή πολλές φορές ανήγγειλε το ξεκίνημα διαπραγματεύσεων για επενδύσεις με το Χονγκ και την Βαϊβάν, αλλά θεωρεί λυπηρό το ότι δεν ξεκίνησαν τέτοιες διαπραγματεύσεις. Με όλα αυτά, υπόψη, το πρόγραμμα της σημερινή ακοράσης και οι συζητήσεις με τους προσκεκλημένους μας θα καλύψουν μια σειρά διαφορετικών εκκρεμών ζητήματα θα βοηθήσουν να βρούμε τρόπου για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δύο πάνελ θα έχουμε. Το πρώτο πάνελ που θα συζητήσει την παρούσα κατάσταση των διμερών οικονομικών σχέσεων με την Ταϊβάν περιλαμβάνει τον κύριο Πίτερ Μπέρτς, γνωστός ε, στα μέλη της Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με έμφαση στην εμπορική διάσταση, τον κύριο Κριστόφ Μανέ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και καλύψει την πολιτική παράμετρο των σχέσεων και τον κύριο Μπαντ Νίνσεν, διευθυντή τη Energon Taiwan, μιας ε, γερμανική επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Ταϊβάν στον τομέα, στον τομέα των ανεμογεννητριών και που θα μας δώσει μια ενημέρωση από πρώτο χέρι για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητε στην Ταϊβάν. Πρώτα πρώτα δίνω τον κύριο, το λόγο στον κύριο Μπέρτς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή τη σημαντική ακρόαση και στον πρώτο πάνελ κιόλα. Να θυμίσω πώς έχει η κατάσταση. Θα παραθέσω αυτά που είπε ο είπατε εκπρόσωπος ε, στη Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί την πολιτική για μία Κίνα, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με την Ταϊβάν. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας ως την μόνη κυβέρνηση της Κίνας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναπτύξουμε στενότερες σχέσεις με την Ταϊβάν. Η συνεργασία και ο διάλογος με την Ταϊβάν γίνονται εντονότεροι σε διάφορου τομείς. Θα σας πει περισσότερα και ο συνάδελφος από, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σχέση με το Ταϊβάν γιατί σεβόμαστε και την μορφή διακυβέρνηση της χώρας. Οι επενδύσεις στην Ταϊβάν είναι σημαντικές και για τις δύο πλευρές και δείχνουν μια δυναμική προσέγγιση. Οι τρεις βασικοί τομείς, αγαθά υπηρεσίες και επενδύσεις. Έχουμε, έλλειψη, έχουμε έλλειμμα στα αγαθά, αλλά πλεόνασμα στις άλλες δύο δομές, όπως τόνισε ο πρόεδρος, είναι ο 16ος εταίρος μας. Έχουμε έναν 50 δις ευρώ εμπορικό όγκο συναλλαγών, όγκος που αυξάνεται, 9 δις εμπορικό έλλειμμα, ωστόσο, για την Ένωση. Στις υπηρεσίες, το διμερές εμπόριο αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. 20% αυξήθηκε με πλεόνασμα 1,7 δις ευρώ το εμπόδιο στις ε, υπηρεσίες συνολικά είναι 10. 50%, 15% αγαθά, 10 υπηρεσίες. Τα στοιχεία του 17 δείχνουν τις εξελίξεις. Η Ένωση ήταν, όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, ο μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής στην Ταϊβάν, 43% των νέων επενδύσεων το 2017. Σε ό,τι αφορά τα εφιστάμενα στόκ, η Ένωση είναι, έχει 28% του συνολικού αριθμού όγκου των επενδύσεων, 50 δις δηλαδή, περίπου. Οι επενδύσεις Ταϊβάν στην Ένωση, από την άλλη πλευρά, είναι μάλλον χαμηλές, 2% μόνο των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε, θα ακούσετε μάλλον περισσότερα στοιχεία από τους άλλους ομιλητές και από το επιμελητήριο, αλλά θέλω να μιλήσω για τις εμπορικές μας σχέσεις. Έχουμε εμπορικές συζητήσεις με την Ταϊβάν, πρόεδρε. Δημιουργήσαμε μια, ένα καλό πλαίσιο διμερού συνεργασίας με μεγάλο αριθμό συζητήσεων και συνεδριάσεων αλλά και Έχουμε δύο ετήσιες ε, διαβουλεύσεις ε, σε εμπορικά ζητήματα το χρόνο. Έχουμε έναν διάλογο βιομηχανικής πολιτικής μια φορά το χρόνο. Τέσσερις ομάδες εργασίας με την Ταϊβάν για τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τεχνικά, φυτογενομικά, φαρμακευτικά και επενδύσεις που συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο. Και έχουμε και μια ομάδα εργασία για την πνευματική διοκτησία που συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Επίσης έχουμε δύο ενδιάμεσες συνεδριάσεις ε, αναθεώρησης πάλι για εμπορικά ζητήματα. Στο πλαίο αυτό τα εμπόδια στο εμπόριο αντιμετωπίζονται και συζητώνται τακτικά αφορώντας ζητήματα νομοθεσίας για τα, καλο, για τα καλλιδικά, ηλεκτρικά αγαθά υψηλού, υψηλού βολτάζ, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και γενικευμένων προτιμήσεων. η Ταϊβάν δεν είναι ε, μέλος σε πολλά όργανα, σε διεθνή όργανα τυποποίησης, αλλά τα θέματα τυποποίησης είναι σημαντικά για μας. Επίσης, η Ένωση με την Ταϊβάν έχουν πρόκειται να ξεκινήσουν ένα νέο φόρουμ ψηφιακής οικονομίας και ενεργειακής συνεργασίας. Υπάρχουν βέβαια τομείς που θα μπορούσαν να έχουμε, θα μπορούσαν να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία. Ενέργεια, Φερρυπίν, ένας από τους καλύτερους τομείς ε, συνεργασίας στην Ταϊβάνια και οι επιχειρήσεις της ε, Ένωσης έχουν μεγάλο πλεονέκτημα στον τομέα των ανεμογεννητριών. Ε, ταυτόχρονα και η γεωργία μπορεί να έχει θετική ανάπτυξη. Τα αιτήματα αδειοδοτηση απο από κράτη-μέλη για μια σειρά προϊόντων, γεωργικό, βόηο, χείριο, ε, πουλερικά κλπ. απορρίπτονται. Προ το παρόν ωστόσο, οι υποχρεώσει πρόσβαση στην αγορά που δεν έχουν υλοποιηθεί δεν είναι πολύ μεγάλες. Εμείς βλέπουμε μεγάλε δυνατότητες στην αύξηση του εμπορίου στον τομέα των βιολογικών προϊόντων αφού η η Ταϊβάν εγκρίνει μια σειρά προδιαγραφών βιολογικών προϊόντων. Τώρα, κρατικές, ε, υπάρχουν και πολλές δυνατότητες κρατικών επενδύσεων, αλλά υπάρχουν και εμπόδια σε αυτό. Υποβολή, υποβολής ε, ε, προτάσεων, έλλειψη εγγράφων στα αγγλικά κλπ. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις εμπορικής συμφωνίας, όπως σας είπα, στην ε, ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου του 2015 για το εμπόριο με όλους, εκφράσαμε την επιθυμία μας η Ένωση να διερευνήσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για επενδύσεις με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Δεν αναγγείλαμε ότι θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, αλλά θα διερευνήσουμε το ενδεχόμενο. Και όντως αναλάβαμε αυτή την δέσμευση και ξεκινήσαμε τις επαφές μας με, τις, με τους φίλους στην Ταϊβάν. Πιο συγκεκριμένα μετά την δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ε, του 2015, η Ταϊβάν και η Ένωση δημιούργησαν μια κοινή ομάδα εργασίας για τις επενδύσεις που συναντήθηκε πέντε φορές μέχρι τώρα. Το 2017, το 2018 και φέτος περισσότερες, στο μέλλον μπορεί να γίνουν περισσότερες συναντήσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε καλύτερη κατανόηση ημέν των επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΔΕ που έχει σημασία λόγω των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε τις εμπορικές διμερείς μας σχέσεις. Προσβλέπω λοιπόν στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών μας σχέσεων και ιδίως σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κριστόφ Μανέ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά λαμβάνω και εγώ μέρο σε αυτή τη δημόσια ακρόαση τη Επιτροπή σα για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Ταϊβάν και ιδίω για τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Το χαιρετίζουμε αυτό. Η Ταϊβάν δεν είναι πάντα το ευκολότερο ζήτημα προ συζήτηση γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνει πολλά ευαίσθητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Κίνας και που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις που έχουμε εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα. Η Ταϊβάν ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα το οποίο παρακολουθείται πάρα πολύ προσεκτικά και από εμά και από την Κίνα και ουσιαστικά ζυγίζουμε πάρα πολύ καλά την κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εδώ πέρα τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Ταϊβάν και να εστιάσουμε περισσότερο στην θετική αξία των επαφών, των εμπορικών που έχουμε. Να δώσω το γενικότερο υπόβαθρο και τη γενικότερη προσέγγιση που έχουμε στη σχέση με την Ταϊβάν και εν συνεχεία θα ήθελα να πω πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι η προσέγγισή μας απέναντι στην Ταϊβάν ουσιαστικά γίνεται σε ένα υπόβαθρο ε, συζητήσεων που έχουν ε, τελματώσει ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν. Όπως ξέρετε, η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοινώθηκε το 2016 προβλέπει μια ευάνθυνση της οικονομικής διπλωματίας και έναν αυξημένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια στην Ασία. Στα πλαίσια λοιπόν του υπόβαθρου αυτού όσον αφορά την ειρήνη και όσον αφορά τη σχέση Ταϊβάν και Κίνας, εμείς θεωρούμε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα αποτελούν προϋποθέσεις όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ασίας και της περιοχής των στενών ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν. Προβλέπουμε ή μάλλον ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μία βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν και ότι θα ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το διάλογο αυτό. Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα αυτό ο διάλογο και λυπούμεθα που οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν έχουν παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Εμείς ε, ανέκαθεν προσπαθούσαμε να πείσουμε και τις δύο πλευρές ε, να έχουν ε, επικοδομητική στάση η μία πέντη στην άλλη και να ξεκινήσουν εκ νέου το διάλογο και προφανώς θέλουμε να υποστηρίξουμε όλες εκείνες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να προωθήσουν το διάλογο, τη συνεργασία καθώς επίσης και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτό και λαμβάνοντα υπόψη και την αυξανόμενη πίεση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, η οποία προσπαθεί να την κάνει να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις διπλωματικές της σχέσεις, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει συγκεκριμένη στρατηγική του 2016 απέναντι στην Κίνα. Το Συμβούλιο προφανώς επιβεβαιώνει την πολιτική για μια ενιαία Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αναπτύσσει περισσότερο τις σχέσεις με την Ταϊβάν και ουσιαστικά να επιμένει περισσότερο στις κοινέ αξίες που διέπουν τις, ε, δύο, τη σχέση των δύο αυτών χωρών και θεωρούμε ότι μπορεί να, να πετύχουμε μια νέα ισορροπία στη σχέση με την Κίνα ερχόμενη σε επαφή με την Ταϊβάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διερευνήσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα περαιτέρω διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν. Και ουσιαστικά αυτή ήταν η στάση που ακολουθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τρία χρόνια και φαίνεται ακόμα περισσότερο τα όσα υπόθηκαν στι 3 Ιανουαρίου από την Επίτροπο Στυλιανίδη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε ο κ. Στυλιανίδη εκπροσωπούσε την κυρία Μογκερίνη. Να σε επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν τότε. Λέμε ότι διατηρούμε προφανώ την πολιτική για μια ενιαία Κίνα, αλλά παράλληλα θα θέλαμε να αναπτύξουμε πιο στενές σχέσεις με την Ταϊβάν, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς που συνάδουν με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και με τους στόχους πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο ακολουθούμε τώρα μια προσέγγιση, ποιο είναι το σκεπτικό. Είμαστε υπέρ του συστήματος διακυβέρνησης που προβλέπεται αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, συγκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊβάν τα τελευταία 30 χρόνια, βλέπουμε ότι η Ταϊβάν έχει δημιουργήσει ένα εμπορικό σύστημα το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένε αξίε, τι οποίε συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Ταϊβάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια προσέγγιση, την ίδια νοοτροπία και ότι ουσιαστικά είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί περισσότερο με την Ταϊβάν, ακόμα και αν δεν υφίσταται διπλωματική αναγνώριση της Ταϊβάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να προωθήσει περισσότερο τη στάση που διατηρεί αυτή τη στιγμή η Ταϊβάν, η οποία αποτελεί πραγματικά υπόδειγμα όσον αφορά το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή τη Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι λοιπόν η συνεργασία και ο διάλογος που έχουμε με την Ταϊβάν γίνονται όλο και πιο έντονοι και συνεχίζουμε να διευρύνουμε το διάλογο αυτό και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε, η γενικότερη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊβάν είναι θετική. Παρ' όλα αυτά, έχουμε επαναλάβει τη δική μας τη στάση σε σχέση με τη θανατική ποινή. Πέρυσι, για πρώτη φορά, είχαμε διαβουλεύσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Ταϊβάν και συζητήσαμε από κοινού όλα αυτά τα ζητήματα. Και το εγχείρημα αυτό ήταν ιδιαίτερα επιτυχές και το φόρουμ αυτό θα συνεχιστεί και φέτος προκειμένου και οι δύο πλευρές να μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες όσον αφορά την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασύνδεση ανάμεσα στο εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υπεράσπιση των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινοτήτων ΛΟΑΔΜΑ, το ζήτημα των συμφερόντων των μεταναστών, το ζήτημα της κατάργησης της θανατικής ποινής και θα συζητήσουμε επίσης και το ζήτημα των εργαζομένων στο βιομηχανικό τομέα. Ήδη υπάρχει ένα ψήφισμα από πέρυσι το Μάρτιο που αναφέρεται στα ζητήματα αυτά και θα συνεχίσουμε το διάλογο αυτό για τα ζητήματα αυτά τον, την Άνοιξη. Η συνεργασία αυτή και όλος αυτός ο διάλογος δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε το εμπορικό και επενδυτικό γραφείο στην Ταϊπέη που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή εκεί, και που προωθεί ιδιαίτερα τις επαφές και το διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν και επίσης διατηρεί τις στενές σχέσεις και αυξάνει, θα έλεγα, τον αριθμό και την ποιότητα των ανταλλαγών απόψεων και σε ζητήματα εκτός του εμπορίου. Ολοκληρώντα, θα ήθελα να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια πιο στενή συνεργασία με την Ταϊβάν, καθότι βλέπουμε ότι συγκλίνουν στην Ταϊβάν και τα συμφέροντα αλλά και οι αξίε μα. Έχοντα αυτό κατά νου, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή ευκαιρία προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πιο θετική δυναμική σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν. Και είναι πολύ σημαντικό η βελτίωση των σχέσεων Κίνας και Ταϊβάν να δημιουργήσει ένα πιο θετικό περιβάλλον για τις περαιτέρω εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ταϊβάν. Θέλουμε η Ταϊβάν να μπορεί να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο σε εξωτερικές σχέσεις. Θα πρέπει η Ταϊβάν να δημιουργήσει περισσότερες σχέσεις με όλους τους διεθνούς παράγοντες και άμεσα με τους ίδιους τους πολίτες και θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα θετικό αφήγημα όσον αφορά την ήπια αυτή δύναμη της Ταϊβάν που θα επιτρέψει την Ταϊβάν να προβληθεί ακόμα περισσότερο και να έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο. Το παράδειγμα της Ταϊβάν είναι θετικό. Θέλουμε να εξελιχθούν θετικά οι σχέσεις με την Κίνα. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τον εμπορικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τα ήδη φυστάμενα εμπορικά εμπόδια, τα οποία θα πρέπει να καταρριφθούν στις σχέσεις εμπορικές που έχει η Ταϊβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Λίνσεν που εκπροσωπεί τη γερμανική εταιρεία Ενερκών. Ευχαριστώ ονομάζομαι Μπαρτλίνσεν και ε, εργάστηκα και ε, έζησα στις, ε, στην Ταϊβάν για 25 χρόνια και έχω χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου, δεν ξέρω τι είναι τώρα πρωί από Εν πάση περιπτώσει, είμαι ο εκτελεστικός διευθυντής της Enercon Ταϊβάν που είναι θηγατρική της ενεργών, της γερμανικής ενεργών ε, που είναι κατασκευάστρια ανεμογεννητριών ε, και επίσης ε, συμμετέχω στην, στην Γερμανο-Ταϊβανέζικη Ένωση Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από το 2005 εργαζόμαστε στην Ταϊβάν και έχουμε συνολικά εγκαταστήσει 230 ανεμογεννήτρες, δηλαδή γύρω στο 70% των νεμογεννητριών της χώρας και έχουμε ε, βέβαια ε, κατακτήσει σχετικές μελέτες ε, για λογαριασμό των ιδιοκτητών αυτών των αεολικών πάρκων. Επίσης έχουμε και ένα περιφερειακό κέντρο διανομής και πωλήσεων αλλά και προμηθειών στην Ταϊβάν και από εκεί και μετά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ταϊβάν είναι υψηλή υπάρχει καταστημένη ε, ικανότητα 50 γιγαβάτ ε, και γύρω στο 50% παράγεται από άνθρακα. Και επίσης ε, η Ταϊπάν διαθέτει το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Και χρησιμοποιείται επίσης και πυρηνική ενέργεια, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκπροσωπούν μόνο το 50% του ενεργειακού μείγματος. Άρα λοιπόν ε, όλες οι, όλα τα ζητήματα απολύσεων και κατανομής της ενέργειας βρίσκονται στο κρατικό μονοπόλιο ε, και η Ταϊβάν έχει θέσει φιλόδοξους ε, στόχους, ε, δηλαδή στο 2025 ε, προβλέπει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας κατά 20% αξιοποιώντας τόσο την νεολική ενέργεια όσο και την, τα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά κυρίως η βιομηχανία εδώ είναι τοπική, παρότι υπάρχουν κάποιε περιορισμένε ευκαιρίε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, ενώ οι, οι κύριες προοπτικές, εδώ απαντούνται για τα ε, υπεράκτια ε, θαλάσσια πάρκα, ε, καθώς προβλέπεται έως το 2000 25 προβλέπεται να κατασταθούν 5 GB συνολικά καταστημένους ισχύω, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν 17 δισεκατομμύρια ε, επενδύσεις, δηλαδή σε ύψος επενδύσεων ε, που θα λάβουν χώρα και ευκαιρίες για, τους, ε, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και βλέπουμε πως κατά τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην Ταϊβάν. Και εδώ αναφέρομαι σε κατασκευαστές αναμογεννητριών, κατασκευαστέ σκαφών, εταιρείε συμβουλευτικές, εταιρείε συντήρησης και εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις ε, που είναι θυγατρικές είτε μεγάλων πολυεθνικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ένα μεγάλο, δύο μεγάλα project έχουν ξεκινήσει ό,τι αφορά τις νέες γεννήτριες. Το ένα τώρα έχει αρχίσει να περάσει στη φάση της υλοποίησης, αλλά τα πράγματα δεν ήταν ε, πάντοτε εύκολα, δηλαδή η ε, διαδικασία της ε, κατακύρωσης ε, περιέλαμβανε μία σειρά από ε, ε, κρατικές υπηρεσίες ενώ υπήρξαν και διάφορες ε, ρυθμιστικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα ενώ υπήρχαν και α, συγκρούσεις αν θέλετε μεταξύ περιφερειακών αρχών που δημιουργήσαν προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Ε, τώρα, η, απαιτήσει σε ό,τι αφορά ε, και το ε, περιεχόμενο αλλά και η ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το, τις δαπάνες ε, των project είναι περαιτέρω προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Εγώ λοιπόν που βρίσκομαι τόσο πολλά χρόνια και εργάζομαι στην Ταϊβάν θεωρώ πως είναι ένας εξαιρετικό χώρο για ανάληψη επιχειρηματική δραστηριότητα με πολύ χαμηλή διαφθορά αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία ακόμα βρίσκεται σε μετάβαση και υπάρχουν δηλαδή κανονιστικά πλαίσια τα οποία δημιουργούν προβλήματα και μπορούν να οδηγήσουν ε, τις ε, ιδιαίτερα τις ξένες επιχειρήσεις σε ε, προβλήματα. Βλέπουμε με βάση την εμπειρία που έχουμε από τους δικούς μας πιλάτες ότι υπήρξαν δημοσίες οι οποίες δεν τηρήθηκαν, υπήρξαν μετακινήσεις για παράδειγμα αεολικών παρκών μετά από πιέσεις που άρχισε η κοινή γνώμη χωρίς να λάβουν αποζημίωση ή υπήρξαν για παράδειγμα αναβολέ ε, σχετικών ε, project για πέντε χρόνια χωρί και πάλι να υπάρξει αποζημίωση. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ορισμένε φορέ έχουμε ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά την, το να λάβουμε έγκριση για ειδικό εξοπλισμό ο οποίο εισάγεται. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο γιατί ε, η Ταϊβάν ε, ορίζει τα δικά τη ε, πρότυπα, πρότυπα δηλαδή τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και στη συνέχεια προστίθεται και μια εγχώρια διάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και εξαρτάται η έκρηση συχνά από τον αρμόδιο τη κρατική υπηρεσία σε, ό,τι αφορά τον ειδικό εξοπλισμό. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα και επιχειρήσει αλλοδαπέ που δραστηριοποιούνται εκεί. Άρα λοιπόν, έχοντα ζήσει 20 χρόνια στην Ταϊβάν, θεωρώ πω είναι πολύ καλεμένο για να ζει ε, καλά μια εύρυθμα λειτουργούσα δημοκρατία, μια ανοιχτή ε, ε, κοινωνία και ε, πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας. Η δική μας εμπειρία στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα καταδεικνύει ότι υπάρχουν ορισμένες, ορισμένα προβλήματα ή δυσκολίες όταν οι στόχοι σε περιφερειακό και σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο διαφέρουν. Παρότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε ό,τι αφορά την τήρηση των στόχων, σε ό,τι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργεια, σε ορισμένε περιπτώσει, ορισμένε αρχέ ακολουθούν τη δική του ατζέντα, τη δική του προτεραιότητα, τη δική του πολιτική. Μία λοιπόν διμερής συμφωνία επενδύσεων θα έδινε τη δυνατότητα και στην ε, κυβέρνηση της ε, Ταϊβάν να επιτύχει ευκολότερα τους δικούς της στόχους για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ε, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εισέλθουν σε αυτή την αγορά, ακολουθώντας τους κανόνες τους οποίους ήδη γνωρίζουν και με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένε στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν εκεί. Εμείς όπω και άλλοι παίκτες εδώ βιομηχανία, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε την Ταϊβάν ω το βασικό ε, κέντρο, αν θέλετε, δραστηριότητά μα για την ευρύτερη περιοχή. Η Ταϊβάν δηλαδή είναι ε, ε, σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της, της ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό λοιπόν στο πλαίσιο και των αιωλικών πάρκων θεωρούμε πω είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει μια τέτοια συμφωνία, διμερή δηλαδή συμφωνία επενδύσεων με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Μάρτιν, ολοκλήρωσαμε τώρα το πρώτο πάνελ. Ερωτήσεις. Ως πρόεδρος, να θέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις για το ξεκίνημα. Πρώτα πάντως στον κύριο Λίντσεν. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που περιγράψετε την δουλειά σας στην Ταϊβάν. Μία ερώτηση μόνο. Είπατε μερικές φορές ότι οι τουρμπίνες κατασκευάζονται και μετά θέλουν τρία χρόνια να συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό είναι λόγω προβλημάτων γενικών ή λόγω μεροληπτικής αντιμετώπισης των ε, ξένων ε, επιχειρήσεων. Δηλαδή υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση όλων ή ευνοϊκότερη των ταϊβανέζικων επιχειρήσεων. Γιατί τους δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπογραμμίστε και οι δύο, δεν ξέρω γιατί, την πολιτική μίας Κίνας. Η πολιτική μίας Κίνας δεν εμποδίζει την Ένωση να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις το μοντέλο του ΠΟΕ μπορεί να μην είναι το καταλληλότερο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις διπλωματικές μας σχέσεις τίποτα δεν υπάρχει που εμποδίζει να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώσουμε διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ταϊβάν είναι μια απόλυτα δημοκρατική χώρα που συμμερίζεται τις αξίες μας Μακάρι να είχαμε τέτοιε και αλλού. Είναι μια χώρα με πραγματική οικονομία της αγορά. Δεν υπάρχει θανατική ποινή, το σωστά είπανε, αλλά υπάρχει στην νομοθεσία πολλών χωρών. Σήμερα ξεκινήσαμε, εγκρίναμε την, ε, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ που εφαρμόζουν την ε, θανατική ποινή. Νομίζω ότι ένας καλός τρόπος ενίσχυσης των σχέσεών μας με την Ταϊβάν είναι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία. Ήδη αναφέρθηκε και θέλω να το ξαναθέσω τι, συμβεί, τι θα συμβεί αν υπογραφεί πριν την υπηρετική Κίνα. Το είπανε κάποιοι, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τέρμα το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων θα έπρεπε να είναι κάτι σημαντικό που θα επιτρέψει να ενισχύσουμε περαιτέρω τους εμπορικού δεσμού που έχουμε με την Ταϊβάν αυτή τη στιγμή. Ας μου απαντήσει κάποιος λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει βέτο από πλευράς Κίνας, για παράδειγμα, ποια είναι η κατάσταση. Η κυρία Αντρικάινεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ του ομιλητές μας. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Μπέρτς, στον Σωστά μιλήσατε για την ε, στρατηγική εμπόριο με όλους του 2015 που πρότεινε η Επιτροπή. Εκεί η Επιτροπή προτείνει να διερευνήσει την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων με το Χονγκ Κόνγκ και την Ταϊβάν. Δυστυχώς, έκτοτε, οι διαπραγματεύσει δεν έγιναν, ούτε καν προτάθηκαν, δεν ξεκίνησαν, ούτε καν προτάθηκαν, ούτε καν αντικτύπου μελέτη αντικτύπου για, ε, για τη διερεύνηση αυτή. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο πριν το τέλος της θητείας της τωρινής επιτροπής. θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Ο κ. Φέρνερ. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε σημαντικό να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις. Δύο ερωτήσεις έχω προς την Κομισιόν μάλλον. Ποιος εξαρτάται περισσότερο από τις καλές εμπορικές σχέσεις, η Ταϊβάνη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, ποιος έχει καλύτερη κατανόηση του τι διακυβεύεται στις, ε, για τις επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ταϊβάν. Αν η Ταϊβάν θεωρεί ότι αυτό θα ήταν χωρίς κίνδυνο, θα συμφωνούσε η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Κρίστοφερ. Σον Κέλλη. Πρώτον, να καλωσορίσω την ευκαιρία τη συζήτηση σήμερα. Ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι. Η υπάρχει πρόθεση και βούληση να βελτιώσουμε την κατάσταση των σχέσεών μας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι ένα διπλωματικό εγχείρημα ή έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε για να δείξουμε ότι θέλουμε πραγματικά καλές εμπορικές σχέσεις με τα Ιβάν το συντομότερο δυνατό. Ποια είναι η θέση της Κίνας θα αντιμετωπίσουμε την Ταϊβάν ως μια ανεξάρτητη οντότητα εμπορικά ή θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Κίνα για να έχουμε μια σαφέστερη θέση. Δεύτερον, <clears throat> άκουσα τι υπόθηκε για την χρήση ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα. Πρόφανώς είναι σαφές ότι Υπάρχει βούληση να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό θα πάρει χρόνο. Έχουν στόχο οι Ταϊβανέζοι ωστόσο για να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα γίνει. Υπάρχουν δυσκολίες στον, προγραμματισμό. Υπάρχουν ωστόσο και τέτοια παραδείγματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρεμποδίστηκαν επιχειρήσεις από κρατικούς ε, ή από, ή από επενδυτέ που να προστατεύσουν τη δική τους επένδυση, εκμεταλλευόμενοι κανόνες σχεδιασμού, το, το χωροταξικού σχεδιασμού που μπορούν να είναι γνωστότεροι στους ντόπιου. Αυτά τα ξέρουμε. Το σημαντικό μήνυμα από την σημερινή συνάντηση είναι νομίζω ότι έχουμε την προθυμία, είμαστε αρκετά θαραλέοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε το σύντομο του δεπτό εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν και να δεσμευτούμε σε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπάλιν, ευχαριστώ πολύ. Απευθύνομαι τώρα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Μπορείτε να μου πείτε αν η Κίνα προσπάθησε να παρέμβει με τον άλλο τρόπο. Γιατί ξέρουμε ότι όσον αφορά τι αερογραμμέ, για παράδειγμα, τι αεροπορικέ υπηρεσίε, ουσιαστικά δεν του επέτρεψαν να μπορούν να έχουν πτήσει προ την Ταϊπέη. Ανάλογη παρέμβαση έχει γίνει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή προς την ΕΙΕΔ από την Κίνα, δηλαδή σας έχουν προτρέψει να μην ξεκινήσετε διαπραγματεύσει συνομιλίε με την Ταϊβάν με τον έναν τον άλλο τρόπο, πρόεδρο. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο οι ερωτήσει. Σα προτείνω να ακούσουμε πρώτα τον Πίτερ, μετά τον κύριο Λίντσεν και τελευταίο τον κύριο Μανέ. Ο Πίτερ πρώτο γιατί είναι πολύ άσχολο, έχει πολλέ ανηλυμένε υποχρεώσει πρέπει να παραστεί και σε κάποιες συνομιλίες που έχει με τους διαπραγματευτές από τη Νέα Ζηλανδία, άρα πρέπει να αποχωρήσει πρώτος. Πίτερ, έχεις πρώτος το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και βέβαια ο συνάδελφο Κριστόφ θα σα δώσει περισσότερε πληροφορίε όσον αφορά την πολιτική που ακολουθούμε. Καταρχά, όσον αφορά τι ερωτήσει σα, καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον που έχετε για το ζήτημα αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Ορισμένες ερωτήσεις είχαν να κάνουν με την επιρροή της υπηρετικής Κίνας, ποια είναι η στάση εμείς απέναντί της και πόσο επηρεάζονται οι πραγματεύσεις αυτές από την πυρωτική Κίνα. Αναφέρθηκα σε ένα επίσημο έγγραφο της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015, όπου λέγεται ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλακεί διαπραγματεύσει με τα Ιβάν. Αυτό λέγεται ξεκάθαρα. Καταρτίζεται όμω έτσι η εμπορική μα πολιτική, όχι προφανώ, αποφασίζεται εδώ στι Βρυξέλλε με τη συμμετοχή Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπή. Και βέβαια η πολιτική για μια ενιαία Κίνα και διορθώστε με αν κάνω λάθο, δεν μα εμποδίζει να ξεκινήσουμε εμπορικέ διαπραγματεύσει με την Ταϊβάν. Η αυτή έγινε πριν από μερικά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο, το, για λόγο δεν ξεκίνησε πραγματεύσει, για ποιο λόγο δεν έγιναν μη τι άλλο μία μελέτη αντικτύπου, για ποιο λόγο βρισκόμαστε ακόμα στη διερευνητική φάση. Κοιτάξτε, για να εξελιχθούν οι πραγματεύσει απαιτείται εντολή. Εντολή προποθέτει πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάση μελέτη αντικτύπου, όπω πολύ σωστά είπατε. Επομένω, η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από το συλλογικό σώμα των επιτρόπων και εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Τι είδου συμφωνία θέλουμε καταρχά Πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την Ταϊβάν, να δούμε ακριβώς τι θέλει κάθε πλευρά και είναι ουσιαστικά ένα διερευνητικό έγγραφο το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε τελικά πού θέλουμε να καταλήξουμε. Έχει όμως η φάση αυτή πολύ μεγάλη σημασία για τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στην πολιτική που θα έχουμε με την Ταϊβάν, στη συνεργασία που θα έχουμε με την Ταϊβάν και θέλουμε να δούμε επίση και ποια είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών. Και η απόφαση του Δικαστηρίου του 2017 ουσιαστικά καθορίζει τη μελλοντική μορφή που θα έχουν οι εμπορικέ μα συμφωνίε και βέβαια οι επενδυτικέ μα μάλλον συμφωνίε, αλλά βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί στην πράξη και δεν έχουμε ακόμα μια τέτοια επενδυτική συμφωνία. Ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή εγκριθεί η συμφωνία με την Σιγκαπούρη και χάρη στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα τα πράγματα κινήθηκαν περισσότερο. Θα έχουμε μία μελλοντική έτσι, πολιτική, εμπορική και επενδυτική. Αυτή είναι μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση τώρα έχει να κάνει με την διαμόρφωση των οργάνων αυτών των δικαστικών για την επίλυση των διαφορών. Πάλι εδώ πέρα κρεμή απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την ΣΥΤΑ και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων το οποίο θα προβλέπεται από τη ΣΥΤΑ και όταν αυτό συνάδει με το νοσιακό δίκαιο. Περιμένουμε εκεί ακόμα να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Και τρίτον, πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσει που έχουμε ξεκινήσει με την πυροτική Κίνα, οι οποίε κινούνται πολύ αργά, αλλά έχουν βέβαια ξεκινήσει, και θέλουμε να δούμε πώ θα εξελιχθούν και οι σχέσει μεταξύ πυρωτική Κίνα και Ταϊβάν. Ίσως τώρα εσείς να θέλετε να συμπληρώσετε κάποια πράγματα, Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να επαναλάβω απλώς ότι όντως η πολιτική για την ενιαία Κίνα δεν μας εμποδίζει να ξεκινήσουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν και άλλωστε αυτό προβλέπεται στα πλαίσια της δικής μας στρατηγικής, στο σχετικό έγγραφο στρατηγικής εμπορικής πολιτικής, όπως ήδη υπόθηκε. Στρατηγική δηλαδή όσον αφορά την Κίνα και όσον αφορά την ε, εμπορική μας στάση απέναντι στην Κίνα. Πολύ ωραία, Στα σύντομο. Κύριε Λίνσεν, εσείς έχετε το λόγο τώρα. Όσον αφορά το ερώτημά σας που έχει να κάνει με την μεροληπτική στάση απέναντι στις τοπικές επιχειρήσεις. Εγώ δέποτε εντόπισα κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η αγορά είναι αρκετά ισότιμη, δίκαιη και ανοιχτή. Οι καθυστερήσεις, στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, έχουν να κάνουν κυρίως με κάποιες περιπλοκές που υπάρχουν στην όλη διαδικασία αδειοδότησης και με κάποιες, θέλετε, τοπικές κυβερνήσεις που δεν συμφωνούν με την πολιτική που επιβάλλεται από την κεντρική κυβέρνηση. Στο μόνο τομέα που θα έλεγα ότι μειονεκτούν κάπως οι ξένες επιχειρήσεις σε σχέση με τις τοπικές είναι ε, το ζήτημα της ενέργειας, κατανομής ενέργειας, δίκτυο το οποίο παραμένει ακόμα κρατικό. Αν έχετε εσείς μια θηγατρική εταιρεία θα πρέπει οποιοδήποτε σύμβαση να διαπραγματεύεται και να υπογράφεται στα Κινέζικα και αυτό αποτελεί μια περαιτέρω επιπλοκή για μα. Σα ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε έτσι τη συζήτηση του πρώτου πάνελ. Α, συγγνώμη, τι το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που έχουμε τελευταία στιγμή και αυτό το λόγο. Ήθελα να θέσω κι εγώ κάποιε ερωτήσει όπω οι συνάδελφοι. Με ικανοποίηση η απάντηση του εκπροσώπου της Επιτροπής στην ερώτηση της κύριε είναι και του κύριου Κέλλη για το timing. Αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το εμπόριο για όλους ότι εκεί προβλεπόταν μια επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν και είναι εύλογο να λέμε ότι με τον ίδιο τρόπο που η που είναι εταίρος ε, με 130 τόσες χώρες και δεν ρωτάει την άποψή μα ε, για την σύναψη συμφωνιών με τις χώρες εκείνες, ομοίως και εμείς δεν χρειάζεται να ζητάμε την άποψη τη Κίνας για την ε, θέσπιση μια συμφωνία. Ε, πέραν αυτού, υπάρχουν, έχουν περάσει πέντε χρόνια σχεδόν από την ανακοίνωση. Είναι και θέμα αξιοπιστία μας. Θα έπρεπε να προχωρήσουμε για να πάρει εντολή κομισιόν ξέρουμε τι χρόνο τρώει 20 χρόνια είναι συμφωνία με το, συζητιέται η συμφωνία με το Μερκοσούρ ε, καιρός είναι να αναλάβουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε υποσχεθεί είναι ένα θετικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα προβλήματα που έχει όπως τη θανατική ποινή. Εγώ άκουσα πολλού συναδέλφους να τονίζουν και συμφωνώ μαζί τους ότι καιρό είναι να πάρουμε μπρο, να προχωρήσουμε με επιφυλακτικό τρόπο ε, ε, εκτιμώντας κάθε παράμετρο της, ε, των διαπραγματεύσεων αυτών αλλά προς όφελος των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης. Εγώ πάντα τονίζω, λέω μπράβο στην Επιτροπή για, την, ε, ε για τις επιτυχίες της εμπορικές της δράσης, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί και τις προτεραιότητες που θέτουν τα νομοθετικά όργανα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος ήθελε το λόγο? Όχι αλλά ούτε και η Κομισιόν θέλει να απαντήσει, γιατί στην ουσία σχόλιο ήταν την ερώτηση. Δεύτερο πάνελ. Που είναι οι προοπτικέ για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένη μια δυνητική διμερού ε, Συμφωνία Επενδύσεων. Καταρχήν έχουμε την ε, κυρία ε, Γιάννη Γιάνγκ που είναι η Γενική Διευθύντρια του ε, Γραφείου Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά έχουμε τον Φρέγκη Χούγκλουντ, ο οποίο είναι ο CEO του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ταϊβάν και θα παρουσιάσει την οπτική γωνία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ταϊβάν. Και μετά έχουμε τον κύριο Τσεν Χουιού από την πολύ γνωστή Ακαδημία σύννεκα τη ε, Ταϊπέη και την παρουσίασε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την ε, Γενική Γιάνκ για την παρουσία τη σήμερα εδώ και τη δίνω κατευθείαν το λόγο. Uh, uh, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι ένας από τους ομιλητές της σημερινής ακρόασης. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το εμπόριο, δεν νομίζω πως χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα ήδη αναφέρθηκαν. Απλώς ε, θα ήθελα να ε, τονίσω τρία σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 51 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το τελευταίο έτος, με αύξηση κατά 8%. Και μάλιστα μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα η, η, η αύξηση αυτή, ή, μάλλον οι εμπορικές συναλλαγές που έχουμε για παράδειγμα σε χοιρινό κρέος, σε βοδινό κρέος ε, και ούτω καθεξούς. Ε, για παράδειγμα είχαμε 45 εκατομμύρια ευρώ σε, σε εισαγωγέ ε, σε ό,τι αφορά το χοιρινό κρέο και είχαμε εισαγωγέ τόσο από την Ισπανία όσο και από την Ιταλία που έφτασε σε 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, το ζαβόν ε, του ε, προσούτου, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ σημαντικό ε, είδο. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τον εμπορικό διάλογο. Από το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ιβάν ξεκίνησαν έναν βιομηχανικό, όπω λέγεται, διάλογο, που εστιάζει στα ρυθμιστικά πλαίσια και στα ζητήματα πολιτική σε ό,τι αφορά την έξυπνη μεταποίηση, την παραγωγή μετάλλων, την μηχανολογία και ούτω καθεξής. Και θεωρούμε πως αυτή η συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική για, ειδικότερα για τις ε, επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές και τις ευρωπαϊκές και τις ΤΕΦΑΝ έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε ε, ε, νέα ζητήματα, νέες προοπτικές. Τώρα, θα ήθελα στο δεύτερο τμήμα της παρέμβασής μου να εστιάσω στις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι εξαιρετικές Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προβαίνει στις υψηλότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην ε, Ταϊβάν ε, φτάνοντας γύρω στα 45 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Δηλαδή αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ταϊβάν. Ε, επίσης, Ε, ε, εγκαταστήθηκε ε, μια, ένα αιωλικό πάρκο με συνολική παραγωγή 5,5 GW που θα πρόκειται δηλαδή για τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αιωλικής ενέργειας στην Ασία και έχουμε εδώ συμμετέχονται στην κοινοπραξία και από τη Γερμανία και από άλλους. Άρα λοιπόν η συνολική επένδυση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά οι στατιστικές ε, δεν ε, ε, αντικατοπτρίζουν τις επενδύσεις τις οποίες προβλέπει η Ταϊβάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι επιχειρήσει δικέ μα συχνά, πολύ συχνά προβαίνουν σε αυτέ τι επενδύσει μέσω τρίτων χωρών. Πάντω, από το, το 2018, με βάση το Σχετικό Ινστιτούτο που έκανε τι σχετικέ έρευνε, διαπίστωσε από το 2008 έω το 2016 οι ταϊβανέζικε επιχειρήσει ε, δημιούργησαν 16.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας λοιπόν ουσιαστικά στην ε, οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ένωσης. Ε, και θα ήθελα εδώ να τονίσω την πρόσφατη ε, εμπορική ε, δυναμική ε, και την διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αντιθέτως δηλαδή προς αυτό η, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος καθίσταται ως ένα και πιο ελκυστικός τόπος επενδύσεων από την πλευρά των ταβανέζικων επιχειρήσεων σε μία σειρά από κλάδους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ε, ε, ψηφίσει ε, τρία ψηφίσματα για τη στενότερη εμπορική συνεργασία μεταξύ Ταϊβάν και Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουμε θερμά αυτή την προσέγγιση του. Από το 2017, όπως ήδη ανέφερε ο Πίτερ, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας και ε, έχει συνεδριάσει πέντε φορές και εγώ είχα συμπροεδρεύσει ενώ συζητήθηκαν μία σειρά από επενδυτικά ζητήματα και θεωρήσαμε πως αυτές οι συναντήσεις ήταν πολύ χρήσιμες και ενημερωτικέ και οι δύο δηλαδή μοιραστήκαμε ε, ε, την πρόοδο που έχουμε επιτύχει σε ό,τι αφορά και τις διαπραγματεύσεις μας και ε, αναφερθήκαμε ειδικότερα στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελευθερού εμπορίου με την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Και βέβαια ε, αναφερθήκαμε και στο, ε, στην πρωτοβουλία που έχει γίνει και από την πλευρά και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ένα πολυμερέ εμπορικό σύστημα. Τώρα, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω από δική μου πλευρά το γιατί χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Ε, θεωρώ πω Ε, ε, ε, θα μπορούσαμε να παράσουμε αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη δικλίδα ασφαλείας για τους επενδυτές γιατί συχνά περιλαμβάνει και προστασία και προώθηση των σχετικών επενδύσεων σε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον και με μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, επειδή ακριβώς δεν έχουν ε, κάποιο άλλο είδος ασθενής συνεργασίας, καλό θα ήταν να αναπτύξουν αυτή τη συνεργασία στο μέλλον. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ταβάνα έχουν τις ίδιες ε, είναι πολύ, ε, βρίσκονται πολύ κοντά μια στην άλλη. Ε, καταρχήν σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις βασικές τους αρχές, σε ό,τι αφορά την ελευθερία, την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία. ενώ σε ό,τι αφορά το εμπόριο και οι δύο πλευρές είναι, επιθυμούν διακαώς να υπάρχει ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα και ένα σύστημα ελεύθερων οικονομιών, το οποίο θα βασίζεται στη διαφάνεια και, στην, και στο σεβασμό του ελεύθερου εμπορίου για όλους. Άρα λοιπόν Είμαστε υπέρ μια τέτοια αυξημένη ε, συνεργασία, αλλά και υπέρ του να ευθυγραμμίσουμε τα δικά μα επενδυτικά εργαλεία περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα. Για παράδειγμα, δεν ε, περιλαμβανόμαστε, δεν συμμετέχουμε σε ορισμένε ομάδε ε, συντονισμού σε ό,τι αφορά αυτέ τι επενδύσει. Για παράδειγμα, οργανώσει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, άρα λοιπόν ε, θεωρώ πως είναι ξεκάθαρα τα ωφέλη ε, και για τις δύο πλευρές από μια τέτοια συμφωνία, ειδικότερα αφού έχουμε πολλές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές οι οποίες προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αιωλικής ενέργειας στην Ταϊβάν. Επίσης, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα ενίσχυε τις διμερείς σχέσεις και θα μπορούσε να ενισχύσει τώρα ε, τι ε, διασυνδέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευρύτερη ε, περιοχή τη Ασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έχει εκφράσει απέναντι σε μια τέτοια δυνητική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν και είμαι βέβαιο ότι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξή σα και στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Χούγκλαντ, ο οποίο είναι επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ταϊβάν. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σα και την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο στην Επιτροπή σα. Εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ταϊβάν, το ECCT, και είμαστε ο βασικό οργανισμό ο οποίο εκπροσωπεί τι ευρωπαϊκέ επιχειρησίε στην Ταϊβάν. Πριν από 31 χρόνια ιδρύθηκε το εμπορικό αυτό επιμελητήριο, από τα παλιότερα στον κόσμο. 400 επιχειρήσει είναι τα μέλη μα και περίπου 900 άτομα συμμετέχουν στο ε, επιμελητήριο αυτό. Όπως είπαν και οι προαλήσαντες, οι Ευρωπαίοι είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Ταϊβάν με 46 δισεκατομμύρια να έχουν επιδηθεί στη χώρα αυτή μόνο και μόνο το 2017. Η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι επένδυσαν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο 64% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ταϊβάν. Τα υπεράκτια ολικά πάρκα αντιστοιχούν σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία επενδύθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσει αυτέ θα πρέπει να προστατευθούν από τι αλλαγέ στο γεωπολιτικό περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο το ECCT υποστηρίζει την δημιουργία μια διμερούς επενδυτική συμφωνία. Μια τέτοια συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να διαφυλάξουμε τι υφιστάμενε επενδύσει. Δεύτερον, να καταφέρουμε να κάνουμε το επενδυτικό περιβάλλον πιο ελκυστικό για τι μελλοντικέ επενδύσει τόσο στην Ταϊβάν όσο και στην Ευρώπη. Πολλέ επενδύσει έχουν τη μορφή κοινοπραξιών και εταιρικών σχέσεων με Ταϊβανέζου επενδυτέ. Πολλοί θα εξακολουθήσουν να επενδύουν στην Ταϊβάν στα πλαίσια πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο τους Ευρωπαίους επενδυτές, αλλά και του εταίρου και του πελάτε του και του προμηθευτέ του σε διάφορε χώρε. Η Ταϊβάν αποτελεί βάση σταθερότητα στην Ασία για πολλέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Τον να επενδύει λοιπόν στην Ταϊβάν κανεί συνάδει με κάποιε πολύ θετικέ επενδυτικέ ευκαιρίε που υπάρχουν, καθότι η Ταϊβάν είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη και σταθερή από την υπόλοιπη περιοχή. Η Ταϊβάν έχει πολύ καλή υποδομή, καθώς επίσης και πολύ καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Είναι ο αγαπημένο προορισμός για διάφορους αποσπασμένους εργαζόμενους και έχει ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο. Ισταρικά όμως η Ταϊβάν έχει καλύτερες σχέσεις και περισσότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πολλοί Ταϊβανέζοι σπουδάζουν εκεί και οι επενδυτέ από την Ταϊβάν πολλέ φορέ αντιμετωπίσουν δυσκολίε με το εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη, με τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Μόνο 13 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμφωνίε αποφυγή διπλή φορολόγηση με Ταϊβάν και για πάνω από 30 χρόνια οι αρχέ τη Ταϊβάν ακολουθούν όλο και περισσότερο διεθνή πρότυπα και βέλτιστε πρακτικέ. Η τάση αυτή συνεχίζεται και τα τελευταία χρόνια. Ως επιχειρηματίες είμαστε ανοιχτοί σε πρακτικούς τρόπους προκειμένου να επιταχυνθεί η τάση αυτή και να επιλύσουμε επιχειρησιακά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές η Ταϊβάν αποκλίνει από τα διεθνή πρότυπα. Πέρα από τα, τις εκθέσει εκθέσεις μας και το διάλογο που έχουμε με την κυβέρνηση, το 2008 δημοσιεύσαμε την πρώτη μας έκθεση που κάνει συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις διμερείς εμπορικές σχέσεις ε, της Ταϊβάν. Επικαιροποιήθηκε η έκθεση αυτή του 2012 και καταδεικνύει τελικά ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα μέτρα αυτά. Την εποχή εκείνη στόχος μας ήταν να προωθήσουμε ουσιώδεις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα βοηθούσαν να υπερκεράσουμε τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια. Από τότε λοιπόν που δημοσιεύθηκε η πρώτη μας αυτή έκθεση, έχουμε συνεχίσει να λέμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία η οποία θα καταφέρει τελικά να ενισχύσει τι εμπορικέ και παιδικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν και που θα βοηθήσει στο να ξεπεράσουμε τα μη δεσμολογικά εμπόδια. Γι' αυτό το λόγο από τότε που ξεκίνησε όλη η συζήτηση για μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν, εμεί την υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν οι εμπορικέ και επενδυτικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για του Ευρωπαίου και Ταϊβανέζου επενδυτέ. Επίση, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τα εμπόδια και το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και επίση θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Θα μπορούσε όμω μια τέτοια διμερή επενδυτική συμφωνία να αντιμετωπίσει και τα εμπορικά εμπόδια. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για την οικονομική ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην Ευρώπη. Τώρα, κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια διμερή επενδυτική συμφωνία. Για παράδειγμα, αν δούμε την σφαιρική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά, την ΣΥΤΑ, καθώ επίση και την επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σιγκαπούρη, βλέπουμε ότι και οι δύο συμφωνίε μπορούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευση για μια μελλοντική διμερή επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Ιδίω όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, ιδίω όσον αφορά τι επενδύσει και ιδίω όσον αφορά το άρθρο 8 τη συμφωνία ΣΥΤΑ, που προβλέπει ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά το νομικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, χώρας εταίρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες που έχουν οι Ευρωπαίοι επενδυτές όσον αφορά τις άμεσες ή ε, έμεσες απαλωτριώσεις που μπορούν να γίνουν στην Ταϊβάν. Το ίδιο ισχύει και για τις ζημίες, καθώς επίσης και την νομική μεταφορά των ε, περιουσιακών στοιχείων. Θα μπορούσαμε να είχαμε διατάξεις όμως για την επίλυση των διαφορών, ιδίως διατάξεις όσον αφορά το σύστημα διαιτησίας μεταξύ επενδυτών και άλλων μερών. Επίση, θα πρέπει να έχουμε κάποιου κανόνε και διαδικασίε για τη διαιτησία, ένα κώδικα διοντολογία για του φορεί διαιτησία και για του διαμεσολαβητέ, καθώ επίση και την εξαρτησία των δικαστικών οργάνων. Επίση, θα πρέπει να γίνει στη συμφωνία αυτή μία αναφορά και στο όλο κόστο κόστος το οποίο θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συμφωνία, καθώ επίσης και σε ένα σύστημα αποζημίωση. Είναι σημαντικό επίση στα πλαίσια μια τέτοια συμφωνία να έχουμε το σύστημα ISDS, την επίλυση δηλαδή διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους και να καταφέρουμε μέσω του συστήματος αυτού να αποφύγουμε οποιαδήποτε πρακτική εισαγωγής διακριτικής μεταχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διευθετήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά, καθώ επίση και με τα μέτρα υγειονομική και φυτογειονομική προστασία για τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ότι όντω υπάρχουν πολλέ μορφέ κρέατο, φρούτων και λαχανικών που εισάγονται από την Ταϊβάν και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαν όμως να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση αν καταφέρουμε να καταρρύψουμε κάποια εμπόδια. Για παράδειγμα, μια αίτηση που είχε γίνει για εισαγωγέ Βρετανικού χείριου κρέατος και είχε υποβληθεί το 2004, εγκρίθηκε το 2018 μετά από 14 χρόνια, ενώ εκκρεμεί ακόμα για 18 ολοκληρά χρόνια μια ανάλογη αίτηση που είχε υποβληθεί για την εξαγωγή ε, βόηου κρέατος από την Ιταλία προς, την Ταϊβάν. Αν καταφέρουμε λοιπόν να εγκρίνουμε μια παιδευτική συμφωνία, θα καταφέρουμε να μειώσουμε και το κόστος αυτό το οποίο εν τέλει μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Τώρα, όσον αφορά τα πρότυπα για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, υπάρχουν πάρα πολλές τοπικές ρυθμίσεις ασφάλειας για την αυτοκινητοβιομηχανία με αποτέλεσμα να απαιτείται διπλή πιστοποίηση και ιδιαίτερα υψηλό διοικητικό άχθος. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να ανοίξουν περισσότερες επενδυτικές ε, ευκαιρίες και να μπορούν και ξένα εργαστήρια να εγκαθίστανται στην Ταϊβάν. Επίση, προβλέπονται συγκεκριμένε απαιτήσει όσον αφορά τι επιδόσεις. Ακούσαμε αυτή τη στιγμή διάφορε παρεμβάσει που έχουν να κάνουν με τον τομέα τη αιωλική ενέργεια. Και εκεί όμω υπάρχουν προβλήματα και εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερκεραστούν για να ευνοήσουμε περισσότερο του Ευρωπαίου επενδυτέ. Πιστεύω επίση ότι όσον αφορά την, τους διαγωνισμούς για τι δημόσιε προμήθειε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο τα κινέζικα αλλά και τα αγγλικά. Νομίζω λοιπόν στα πλαίσια μια διμερή επενδυτική συμφωνία θα πρέπει να καλύψουμε πάρα πολύ και τι ανησυχίε των Ευρωπαίων. Ποιε είναι οι ευκαιρίε όμω τώρα για την ίδια την Ευρώπη. Οι ξένε επενδύσει τη Ταϊβάν αυξάνονται όλο και περισσότερο από το 1990. Από το 2006 οι συνολικέ αιτήσει επενδύσει ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω και για πολλά χρόνια από το 2012 και μετά έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρ' αυτά, ελάχιστα από τα χρήματα αυτά καταλήγουν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρώπη μπορούσε να προσελκύσει έστω και ένα μικρό μερίδιο τη εξωτερική επένδυση τη Ταϊβάν, αυτό από μόνο του θα καθιστούσε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη μια τέτοια διμερή επενδυτική συμφωνία. Μια τέτοια συμφωνία επίση θα προέβαλε περισσότερο την Ευρώπη ως προορισμό επενδύσεων από την Ταϊβάν. Επίσης, η Ευρώπη έχει ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας, ενώ η Ταϊβάν από την άλλη χρειάζεται πολύ περισσότερους εργαζόμενους, τόσο ειδικευμένους όσο και ανειδίκευτους. Επίσης, μία αύξηση στις διμερείς επενδύσεις που θα μπορούσε να έρθει μέσω της συμφωνίας αυτής θα μπορούσε να οδηγήσει και σε καλύτερη ανταλλαγή γνώσης και δεξιοτήτων. Εν κατακλείδη, η διμερή επενδυτική συμφωνία μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο ζητάνε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει στην Ταϊβάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η συμφωνία αυτή δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα πρόσβαση στην αγορά, αλλά θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα αποτελέσει κίνητρο για να υπερκεραστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα και ουσιαστικά θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κάποια νέα ζητήματα που έχουν προκύψει, όπω η βιοιατρική, η κυκλική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι λοιπόν να κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τι ευρωπαϊκέ επενδύσει στην Ταϊβάν, ιδίω σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώ. Και νομίζω ότι ο σημαντικότερο λόγο για να έχουμε μια τέτοια διμερή επενδυτική συμφωνία δεν είναι όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στα, στα, στα όσα σα είπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ταϊβάν είναι μια ήπια δύναμη στην ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει πραγματικά να ληφθεί υπόψη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι και από πολιτιστική πλευρά πρέπει να έχουμε μια τέτοια συμφωνία, καθότι θα συμβάλλει στι μακροχρόνιε αυτέ εμπορικέ και επενδυτικέ σχέσει που υφίστανται μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Η καθηγήτρια κυρία Γου και ο καθηγητή κύριο Γου. Είμαι δικηγόρος ο πρώτος Ταϊβανέζος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Η ερώτηση που θέτω στον εαυτό μου είναι η εξής. Γιατί δεν υπάρχει δεν υπάρχουν εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊβάν. Και πάλι, γιατί η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει να μην προχωρήσει σε διάλογο με την Ταϊβάν αντί να προχωρήσει σε πιο σε μέτρα που βασίζονται στο νόμο. Αυτά είναι μια σειρά ερωτημάτων που θέτω. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να σας θυμίσω ότι το άθρο 21 της συνθήκης λέει, του ΑΣΕΑΝ λέει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις με την Ταϊβάν και αυτό μας οδηγεί στην συζήτηση του πώς, μπορούν η, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Ανατολική Ασία προτείνω μια σειρά στρατηγικών για την επένδυση, για τις επενδύσεις. Το πρώτο είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, το δεύτερο μια συμφωνία επενδύσεων και τρίτη νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ταϊβάν. Ήταν κάτι, είναι κάτι πολύ θετικό για μας και αυτό θέλαμε πάντα. Το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η... υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. E Επίσης, μία επιλογή είναι μια συμφωνία επενδύσεων μεταξύ των δύο των δύο πλευρών. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Εμπόδιο και Όλο. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι παρά τις ε, ελπίδες της Ταϊβάν και μια σειρά ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι διαπραγματεύσεις δεν ξεκίνησαν ακόμα. Το πρώτο λοιπόν και πιο σημαντικό καθήκον για μια τέτοια συμφωνία είναι να ξεκινήσουν οι σχετικέ συζητήσει, που σημαίνει η Επιτροπή να ζητήσει εντολή διαπραγματεύση από το Συμβούλιο και να εγκριθεί κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο. Δίνοντας εντολή θα κινητοποιήσει τι διμερείς διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο πλευρών και ταυτόχρονα θα βοηθήσει να τερματιστεί η... το τέλμα στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσης, μια συμφωνία επενδύσεων θα είναι θετική για τις επενδύσεις των δύο πλευρών και αυτό πρέπει να ξεκινήσει κατά συνέπεια. η μελέτη αντικτύπου πρέπει να γίνει αμέσως. Μια τέτοια συμφωνία είναι υπέρ και της Ένωσης και των επιχειρήσεών της. Από την οπτική της Ένωσης θα δώσει μεγαλύτερη επένδυση, μεγαλύτερη υποστήριξη σε ένα, στο σύστημα, επίλυσης των διαφορών επενδύσεων καθώς η Ταϊβάν θα χαρεί ιδιαίτερα να, ένα τέτοιο, να δεχθεί ένα τέτοιο σύστημα και δεν είναι μέλος στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Επιχειρήσεων. Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, οι επενδύσεις ε, σε offshore, σε υπεράκτιες ε, ανεμογεννήτριες θα κερδίσουν σημαντικά. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν και το περιβάλλον θα έχουν δε και σαφή παράμετρο περιβαλλοντική. Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών έχει πολιτικές ε, αμφισβητήσεις. Δηλαδή, ε, υπάρχει ένα ε, ερώτημα. Θα έπρεπε η Ένωση να ξεκινήσει πρώτα μια τρίτη συμφωνία με την Κίνα ή με την Ταϊβάν. Σίγουρα αυτό είναι πολιτική επιλογή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν προηγούμενα σε άλλες αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Μπορούν κάλλιστα οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν παράλληλα. In fact, the EU concluded bilateral WTO accession negotiation with Taiwan first, then with China. So there's no pro there should be no problem for the EU to negotiate simultaneously a BIA with Taiwan. Moreover, in the context of AFSA,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 And sometimes you have to ask questions even though you partly know the answer because you have to get things <laughs> up in the air and out in the open. Uh, we've we signed free trade agreements with Japan. We signed... Έχουμε υπογράψει ε, ε, τέτοια ε, συμφωνία με την Ιαπωνία, το κάναμε με την Κορέα και το κάνουμε μόνο με τα περισσότερες χώρες της περιοχή. Οπότε, αν ήμουν οικονομολόγο από την Ταϊβάν θα με ανησυχούσε αυτή η τάση και πραγματικά δεν νιώθω ικανοποιημένο με αυτό δεν θεωρώ πως είναι δίκαιο με τον τρόπο δηλαδή που ε, διαμορφώνεται η παραγωγή σε αυτήν την περιοχή. Και αν ακούσω και τα όσα μας λέει και το επιμελητήριο, ε, τότε ε, τα όσα προβλήματα μας αναφέρεται και τώρα τα ζητήματα ανησυχία είναι αυτά ακριβώς που αντιμετωπίζουμε μέσω των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Αυτά μας απασχολούν εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Αλλά από τότε που αναφέρεται αυτό το ζήτημα, ουσιαστικά προσπαθούμε να αναβάλουμε έτσι πολύ διακριτικά αυτή τη σύναψη μιας συμφωνίας ε, επενδύσεων ή BIA ή BIT όπως ε, θέλετε να την ονομάσετε. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις ευαισθησίες ε, των άλλων, γι' αυτό νομίζω πως το μαθαίνει κανείς σιγά σιγά, επιβιώνοντας τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ο λόγος για τον οποίο συζητούμε ε, μια συμφωνία επενδύσεων ε, και όχι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι επειδή σέβεστε τις δικές μας ευαισθησίες ή επειδή σέβεστε τις ευαισθησίες του μεγάλου γείτονά σας. Ε, γιατί βέβαια θεωρώ πως εμείς ως αυτόνομη αν θέλετε οικονομική δύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Ε, δεν θα θέλαμε δηλαδή εμεί να κινήσουμε τι διαπραγματεύσει με κάποιον ο οποίο φοβάται να μην βλάψει τα συμφέροντα ενό ε, τρίτου. Άρα λοιπόν ο λόγο για τον οποίο, επαναλαμβάνω, προτιμούμε μια συμφωνία BIA, ε, μάλλον προτιμάτε εσεί μια συμφωνία BIA αντί για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, είμαστε εμεί ή είναι ο μεγάλο γείτονά σα. Ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Γιάνγκ, με εξέπληξε τα, το γεγονός που ο κύριος Χόμπλουν μίλησε για αυτά τα μη δασμολογικά εμπόδια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα αυτό. Επίσης, τι δυνατότητες μεγαλύτερων επενδύσεων από πλευράς Ταϊβάν υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και μια άλλη ερώτηση που μπορώ να τη συζητούμε μακρόν, αλλά θέλω να το κάνω σύντομο, είναι ποιε είναι οι σχέσει μεταξύ Ταϊβάν και υπηρετικής Κίνα αυτή τη στιγμή. Για τον καθηγητή τώρα. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να ξεκινήσουν παράλληλες διαπραγματεύσεις με την υπηρετική Κίνα. Η Κίνα βέβαια δεν είναι δημοκρατία, ενώ η Ταϊβάν είναι. Η ποιοτική Κίνα δεν είναι ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Η Ταϊβάν είναι. Γι' αυτό θεωρώ άδικο υπό τις συνθήκες αυτές να, είμαστε, να μας παρεμποδίζουν ε, οι Κινέζοι να ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αν δεν θέλει η Κίνα, εντάξει, δύσκολο, αλλά θα το πετύχουμε. I think that concludes the questions. I'm going to go back to the panel and then after. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε εδώ τις ε, ερωτήσεις. Ε, να δώσω λοιπόν ε, το λόγο στους ομιλητές του πάνελ και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κ. Τζογκάνη για να ολοκληρώσει. Ε, και θα σας δώσω τον λόγο ε, Πρώτα σε σας ε, κύριε Ρούγκλου και, και στη συνέχεια στους δύο ε, αν δεν ε, θεωρείτε πως καμία ερώτηση απευθυνόταν σε εσάς, τότε δεν χρειάζεται να πάρετε το λόγο. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο μιλτή. Um, again, I, I present, I'm a trade lawyer. Είμαι ε, νομικός επιβολικών συστημάτων και ως νομικός ε, προετοίμασα δύο ε, διαφορετικές εναλλακτικέ στο δικό μου έγγραφο, δηλαδή από τη μία συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου, από την άλλη BIE ή και από την άλλη μια συμφωνια ελεύθερο εμποριου απο την αλλη bie η και απο την αλλη μια συμφωνια για την επίλυση ορισμένων ζητημάτων, όπως για παράδειγμα του κανονισμού προστασία των δεδομένων και ούτω καθεξής. Αλλά όπως είπαμε βέβαια, η πιο, η πιο φιλόδοξη λύση είναι αυτή τη συμφωνία ελεύθερο εμπορίου. Ωστόσο μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα. Δηλαδή, μια συμφωνία ε, επενδύσεων μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ή με μια συμφωνία πιο ε, κλαδική, δηλαδή με συγκεκριμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Άρα λοιπόν, το ερώτημα που θέσατε ουσιαστικά βρίσκει μια απάντηση από την δική μα πλευρά, δηλαδή από μένα ω νομικό, ε, στην ισορροπία που προσπαθώ να βρω ανάμεσα στην φιλοδοξία αφενό και το τι είναι δυνατό, τι είναι ρεαλιστικό να εφαρμοστεί. Και στο έγγραφό μου λοιπόν εγώ ανέλησα το πώς έχουν τα πράγματα εφόσον παραμείνει το status quo ως έχει σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω αν έχετε το έγγραφο διάθεση, αλλά από ό,τι κατάλαβα έχει δανειμηθεί ήδη στα μέλη τη Επιτροπή. Πολύ καλά. Ε, ο λόγο τώρα στην κυρία Αγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά τις ερωτήσεις που έθεσαν ε, οι ευρωβουλευτές, θα ήθελα να πω ότι καταρχάς πριν από 10 χρόνια θέλαμε να δημιουργηθεί μια, να θεσπιστεί μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο όμως δεν έχουμε καταφέρει να συνάψουμε εμεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υφίσταται ουσιαστικά μια ανάλογη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη ή την Ιαπωνία. Το θέμα νομίζω έγκυται περισσότερο στο ότι αν πραγματικά χρειαζόμαστε μια τέτοια FTA, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. θέλουμε εμεί συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθότι δεν συμμετέχουμε σε πάρα πολλού διεθνεί εμπορικού οργανισμού, να καταφέρουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα, να καταφέρουμε να μάθουμε από εσά. Είτε μιλάμε για τα εμπορικά εμπόδια, είτε μιλάμε για ζητήματα υγειονομική, φυτογενομική προστασία καθεξής. Αλλά ήδη από το 2015 και τη σχετική ανακοίνωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο εμπόριο για όλους, είπατε ότι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να ξεκινήσει επενδυτική συμφωνία, επενδυτικές διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν και επαναλήφθηκε η πρόθεση αυτή και το 2018. Εμείς ουσιαστικά συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, FTA, προϋποθέτει και ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής συνεργασίας. Γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε εμεί ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με μια BIA, με μια διμερή επενδυτική συμφωνία, καταφέρνοντας να καλύψουμε κάποια διμερή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και την προώθηση των επενδύσεων. Όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου, προφανώς μια τέτοια συμφωνία θα προωθήσει περισσότερο τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις προς την Ταϊβάν και το αντίστροφο. Νομίζω ότι Μέσω μια τέτοια συμφωνία μπορούμε πάντω και εμεί ω Ταϊβάν να μάθουμε πάρα πολλά από εσά όσον αφορά τι εμπορικέ διαδικασίε. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει για μια διμερή επενδυτική συμφωνία και καταλαβαίνω βέβαια, συνειδητοποιώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έχει συνάψει ακόμα τέτοιες επενδυτικές συμφωνίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εξετάστε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε τέτοιες διαπραγματεύσεις με κάποιες χώρες. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να ξεκινήσουμε σχετικές διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία με εσά, με τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Άντρε Κάιν έχει τώρα το λόγο για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη αξιότιμη ε, προσκεκλημένη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη αυτή ε, συνεισφορά σας στη σημερινή ακρόαση. Θα ήθελα να επενθυμίσω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπέρ διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν για μια επενδυτική συμφωνία βάσει της, του ψηφίσματος του 2018, το οποίο καλεί την έναρξη τέτοιου διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊβάν. Όπως ήδη υπόθηκε πολλές φορές σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές στο παρελθόν πρότεινε να διερευνήσει τη δυνατότητα έναρξης τέτοιων επενδυτικών συμφωνιών με την Ταϊβάν. Δυστυχώς όμως διαπραγματεύσεις αυτές δεν ευωδόθηκαν, δεν ξεκίνησαν καν. Και ένας λόγος τελικά είναι ότι δόθηκε προτεραιότητα σε επενδυτικέ διαπραγματεύσει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας οι οποίες όμως βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει μόνο να επικεντρωθούμε σε επενδυτικέ διαπραγματεύσει με την Ταϊβάν, αλλά θα μπορούσαμε ακόμα και να προωθήσουμε έναν σφαιρικότερο διορθρατικό διάλογο για το εμπόριο, ιδίως μέσω των ομάδων εργασία και άλλων διαρθρωτικών μέσων διαλόγου. Προτείνεται μάλιστα να ξεκινήσουν οι πραγματεύσει αυτές, αλλά απουσία κάποιας μελέτη αντικτύπου έχουν συσταθεί συγκεκριμένε τεχνικέ ομάδε εργασία για ζητήματα όπως τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όσον αφορά τα μέτρα υγειονομικής και φυτονομικής προστασίας, ζητήματα διανοτικής ιδιοκτησίας, φαρμακευτικά ζητήματα και τέλος μια μάδα εργασία για τις επενδύσεις. Στις ε, τομεακές αυτές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της ενέργειας, προωθείται μία τομεακή ε, συνεργασία, η οποία βέβαια δεν φτάνει το επίπεδο φιλοδοξίας που θα μπορούσαμε να είχαμε όπως στα πλαίσια μιας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας, αλλά αποτελούν μία λύση προκειμένου στο και βραχυπρόθεσμα να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊβάν. Όπω άλλωστε είπαν και συμμετέχονται στη συζήτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο θαραλέα και να κινηθεί σε πιο διαθρωμένες εμπορικέ σχέσει με την Ταϊβάν. Όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Χου πριν από λίγο, η εντολή που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει συζητήσει για μια BIA με την Ταϊβάν θα μπορούσαν ουσιαστικά να συμβάλλουν στο να ξεπεράσουμε το διέξοδο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει στι σχετικέ διαπραγματεύσει με την Κίνα. Υπό το φω τη πρακτική που ακολουθείται στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι διαπραγματεύσει με την Κίνα και με την Ταϊβάν θα μπορούσαν να εξελιχθούν παράλληλα. Δεν θα πρέπει να υφίσταται κανένα πρόβλημα στο να καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε παράλληλα με την Κίνα και μια διμερή παιδιτική συμφωνία με την Ταϊβάν. Επίσης υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει θεωρήσεις σε πολίτες της Ταϊβάν χωρίς να έχει την ίδια ευέλικτη προσέγγιση σε πολίτες της Κίνας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κινηθούμε ανεξάρτητα στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν. Τώρα όσον αφορά την μελέτη αντικτύπου. Αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για να οδηγηθούμε σε μια διμερή επιδετική συμφωνία και προτού ολοκληρωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τρέχουσα θητεία, θα θέλαμε πραγματικά να δούμε να ελοποιείται αυτή η μελέτη αντικτύπου. Είναι μια πλήρως αναπτυγμένη δημοκρατία η Ταϊβάν, η οποία συμμερίζεται κοινέ αξίε όπω η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, σεβασμό του κράτου δικαίου, καθώ επίση και μια οικονομία που βασίζεται στι αγορέ. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, μία διμερή επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν θα επεκτείνει τι υφιστάμενε επενδύσει και θα δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο προκειμένου να υπάρχει μια σταθερή νομική προστασία. Μία συμφωνία εμπορική θα μπορούσε να καλύπτει και τον τομέα της πρόσβασης στην αγορά, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να καλυφθούν και άλλοι τομεί όπω υπηρεσίε και βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένα μηχανισμό προστασία των επενδύσεων. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συμμετέχοντε από την Ταϊβάν που ήρθαν σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι χάρη στι κοινέ μα προσπάθειε η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και θα οδηγήσει σε πολλά κοινά ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ε, πολυθετικές με αυτά τα πολύ θετικά συμπεράσματα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές του πάνελ, ειδικότερα εκείνους που προσήλθαν από την Ταϊβάν ε, σήμερα εδώ. Ε, και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που ανέφερε η συγκήτρια, ότι δηλαδή η, δική μας θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι προτού ολοκληρώσουμε τη δική μας θητεία του τρέχοντο Κοινοβουλίου θα θέλαμε τουλάχιστον, τουλάχιστον το ελάχιστο να έχει ολοκληρωθεί η ε, αξιολόγηση αντικτύπου μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώνεται εδώ η ακρόαση.